Καλησπέρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Και καλωσορίσατε στην δεύτερη μας ε, συνάντηση ε, εξ αποστάσεως. Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά είδαμε πώς γίνεται η ψηφοφορία εξ αποστάσεως και σας ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική συνεργασία. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και την ε, γραμματεία που προτίμασε με άριστο τρόπο όλα αυτά. Η σημερινή μας ημέρα διάταξη έχει μόνο την τελική ψηφοφορία για ε, το, τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις για τον προπολισμό της χρήσης του 2021 και το Κοινοβούλιο θα πρέπει έτσι να συνεχίσει και θα πρέπει να ακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή τις οδηγίες. Μετά από όλα αυτά θα μπορούμε να δούμε τι λέει η ημερησία διάταξη. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση τότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Καλώς. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά την ε, διερμηνία. Θα έχουμε προς αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά και πορτογαλικά. Λέει ο αλλά έχουμε και πολωνικά, αντί των πορτογαλικών. Και θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις δεν θα μεταφράζονται, οπότε παρακαλώ ε, όταν λαμβάνετε το, χώρο, να, το λόγο να μιλάτε με φυσιολογικό ρυθμό και έτσι να μπορούν να σας μεταφράσουν οι διερμηνείς όπως πρέπει. Την περασμένη εβδομάδα ψηφίσαμε για τον συμβιβασμό μεταξύ της Επιτροπής μας και του Προεδρείου όσον αφορά τον προπολισμό του 2021. Υπενθυμίζω ότι προβλέπεται αύξηση 2,54 σε σχέση με το 2020 και επίσης καλύφθηκαν και οι τροπολογίες για το σχέδιο κειμένου και σήμερα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία. Πρώτα πρώτα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον έχουμε την απαραίτητη απαρτία ε, που είναι 11 συνάδελφοι παρόντες. To click or tap the race hand. Α, θα πρέπει να σηκωστώ χέρι σας ή να πατήσετε το σχετικό κουμπί. Αυτό το κουμπί βρίσκεται στην οθόνη για την πλατφόρμα της Interactio. Και έτσι να δούμε αν υπάρχει απαραίτητη απαρτία. Όλοι οι συλλαμβάνουμε στην ψηφοφορία έχουν πάρει τη σχετική ε, ε, λίστα ε, σε πρωτόκολλο σε μορφή PDF την Παρασκευή και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι για να είναι έγκυρη η ψήφο σα θα πρέπει να ψηφίσετε μεταξύ 5 και 6 πρώτα πρώτα. Συμπληρώστε αυτό το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο στην ε, οθόνη σας με το πληκτρολόγιο σας. Μετά θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα αντίγραφο ε, του συμπληρωμένου εγγράφου και εκεί υπογράφεται τη σχετική δήλωση. Μπορείτε αυτό να το κάνετε με εκτυπωτή ε, ή με, να το κάνετε με το χέρι σας και μετά να το σκανάρετε ή με αυτό το ειδικό μολυβάκι για τις ε, οθόνες αφής. Και αυτά θα τα στείλετε σε αυτό τη διεύθυνση ε, email που έχετε λάβει, αλλά θα γίνει από τη διάθεση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επίσημη, τη δική σας, του Κοινοβουλίου. Μόλις αρχίσει η ψηφοφορία θα κλείσουμε την συνεδρίαση. Δεν θα ξανασυναντηθούμε για τα αποτελέσματα. Θα στα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οπότε η τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει την 5η ε, 14 σε σχέση με τις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό. Έναρξη της ψηφοφορίας και ταυτόχρονα λήξη της συνεδριάσεως. Και σας ευχαριστώ.